Αυτό που ακολούθησε ήταν ότι δεν υποστηρίχθηκε αυτή η συμφωνία από το Συμβούλιο και μετά από την διοργανική συμφωνία και αφού ξεπεράστηκε το θέμα της κατεξουσιαδότησης πράξης και προχώρησε και το θέμα της, της νομοθεσίας. Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες επεξεργάζονται αυτήν την συμφωνία. Μετά από δύο χρόνια λοιπόν ελπίζω να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και ίσως να ψηφίσουμε τον Απρίλιο στην επόμενη συνεδρίασή μας και να περάσει και από την Ολομέλεια το Μάιο. Εκρεμεί εδώ και πολύ καιρό αυτό το θέμα και ελπίζω να προχωρήσει. Αυτά όσον αφορά το σημείο 7 και να περάσουμε και στο σημείο 8. Και κλεισμένο το θερόν αυτό, αγαπητοί... Α, όχι. Έκανα λάθος. Έτσι λένε οι σημειώσεις μου. Ωραία δημόσια θα συζητηθεί το θέμα αυτό. Μπορείτε να μείνετε όλοι στην αίθουσα. Λοιπόν, πρόκειται για ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με την ε, έκθεση παρακολούθησης για το TTIP. Θυμάστε αυτό το εξαιρετικό ψήφισμα της 8 Ιουλίου ήταν το μήνυμα που θέλαμε να στείλουμε προς τους διαπραγματευτές. Είναι η θέση του Κοινοβουλίου για κάποια συμφέροντα επιθετικά και προστασίας και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε την Επιτροπή. Πώς έχετε επεξεργαστεί αυτό το κείμενο της 8 Ιουλίου. Η Επιτροπή βεβαίως έχει δημοσιεύσει τον Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου του 2015, την έκθεσή της και σήμερα μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για την έκθεση αυτή. καθώς και για την ε, υλοποίηση δική, του δικού μας ψηφίσματος. Στην τελευταία ομάδα παρακολούθησης συζητήσαμε το θέμα αυτό και βεβαίως ήθελα εδώ να καλωσορίσω και τον αναπληρωτή αντιπρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τις Ηνωμένε Πολιτείε και τον Καναδά. Με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενσωμάτωσε τις προτάσεις μας στις διαπραγματεύσεις του Καναδά και της ΗΠΑ. Μία πολύ σύντομη απάντηση θα σας δώσω. Λάβαμε υπόψη την διεξοδική πρόταση ψηφίσματος του Ιουλίου, όπου ήρθατε σε επαφή και με άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου και που σχετιζόταν και με τη δική μας εντολή. Ήταν λοιπόν ένα χρήσιμο συμπλήρωμα στις άλλες ε, κατευθυντήριες γραμμές διαπραγμάτευσης που είχαμε. Η ουσία είναι αυτό ακριβώς που είπατε, δηλαδή να μιλήσουμε για τα επιθετικά και αμυντικά μας μελήματα καθώς και τις κόκκινες γραμμές. Και αυτό που προσπαθήσαμε ήταν να διασφαλίσουμε ότι, ότι θα πρέπει να υπάρξει μία ε, ποιοτική συμφωνία ε, εκτενής και ισορροπημένη. Η Επίτροπος ε, πολλές φορές, σε σχέση με το πρώτο θέμα, σε σχέση δηλαδή με το επίπεδο προστασίας, ότι το TTIP δεν θα μειώσει το προστατευτικό πλέγμα σε καμία πλευρά του Ατλαντικού. Σε σχέση με τον διεξοδικό χαρακτήρα της συμφωνίας, η Επίτροπος Μάλμστρεμ τους, προηγούμενου τους προηγούμενους μήνες ε, ανέφερε ότι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μια ήπια συμφωνία με τις ΕΠΑ, κάτι το οποίο συμμερίζονται και οι ομολογοί μας. Ως προς την εξισορρόπηση δεν θα θέλαμε να προβλέψουμε μια συμφωνία που να είναι φιλόδοξη για τις ΗΠΑ και ε, μετριοπαθής για εμάς. Θα θέλαμε να φτάσουμε σε μια εξισορρόπηση. Τώρα, έμπρακτα, πού βρισκόμαστε Έχουμε 13 προσχέδια ε, κεφαλαίων και προσπαθούμε να φτάσουμε σε ένα ενιαίο κείμενο με αγγίλες εκεί όπου υπάρχουν διαφορές. Και αυτό βρίσκεται μεσοστρατής του κειμένου, του τελικού κειμένου που περιμένουμε στο τέλος της εργασίας. Έχουμε δηλαδή το ίμιση της εργασίας, το ίμιση των κεφαλαίων. Μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα είχαμε ανταλλαγές απόψεων στις δημόσιες προμήθειες και αυτό αφορά το τελικό στάδιο της πρόσβασης στην αγορά μετά από προτάσεις ως προς τους δασμούς και τις υπηρεσίες. Μετά από τις έντονες διαβουλεύσεις για την προστασία των επενδυτών και των επενδύσεων υποβάλαμε μία αναθεώρηση πέρσι τον Μάιο και φτάσαμε σε ένα ενιαίο σύστημα προστασίας των επενδύσεων που υποβάλαμε και στις δύο πλευρές. Και έχουμε αρχίσει να διαπραγματευόμαστε με τις ΕΠΑ για τις ενδεχόμενες ε, παραμέτρους ε, προστασίας των επενδύσεων στο TTIP. Ο τελευταίος γύρος του Φεβρουαρίου οδήγησε σε ανταλλαγή κειμένων σε σχέση με την κανονιστική συνεργασία σε αυτή την ενδιάμεση φάση και εργαζόμαστε και εμείς και η Επίτροπος που ήρθε σε επαφή με τον ομολογό της την προηγούμενη Παρασκευή στις ΕΠΑ. Επίσης, σε σχέση με τις παραμέτρους ε, του ψηφίσματος του Ιουλίου, υποβάλαμε στις ΕΙΠΑ τα Χριστούγεννα μια φιλόδοξη πρόταση για βιώσιμες ε, προτάσεις και την προστασία του περιβάλλοντος. Βρισκόμαστε στο μέσον αυτής της διαπραγμάτευσης θα ενσωματώσουμε τις διάφορες παραμέτρους που διέπουν και τη δική σας ε, πρόταση ψηφίσματος. Ελπίζω μέχρι το καλοκαίρι να καλύψουμε όλες τις πτυχές της διαπραγμάτευσης και ο εκπρόσωπος των ΙΠΑ ζήτησε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με τη λήξη της θητείας της κυβέρνησης Ομπάμα. Και φυσικά το περιεχόμενο υπερέχει όλων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος της Επιτροπής για το ψήφισμά σας και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ενδεχόμενες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα αλλάξω ιδιότητα. Θα θέσω κάποιες ερωτήσεις ως εισηγητής για το θέμα αυτό. Διάβασα την έκθεσή σας προσεκτικά, ε, στην οποία σχολιάζεται το ψήφισμα και έχετε σαφή άποψη για το τι σημαίνει το ψήφισμά μας. Όμως, στις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις θα έλεγα ότι κυριάρχησε η περιγραφή, ήταν κάπως άνευρες. Επομένως πράγματι έχω και πιο συγκεκριμένες ερω... ερωτήσεις να θέσω. Στο ψήφισμά μας για τα γεωργικά είπαμε ξεκάθαρα ότι Θέλουμε να έχουμε ένα αποδεκτό επίπεδο της ε, καλής διαβίωσης των προτύπων για την καλή διαβίωση των ζώων και να είναι ισότιμο με το ε, επίπεδο που επικρατεί ε, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αναφερόμαστε στα προϊόντα που εισάγονται στο ευρωπαϊκό έδαφος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς θα το υλοποιήσετε αυτό το προαπαιτούμενο στις διαπραγματεύσεις. Τώρα για τις οριζόντιες διατάξεις για εξαιρέσεις την ΚΑΤΣ, άρθρο 14. Πώς το συμπεριλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις αυτό. Και τέλος, το θέμα του ωφέλους για τις τρίτες χώρες. Στην έκθεσή σας αναφέρεστε κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς αναγνωρίζετε τις ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών στη διαπραγμάτευση για την TTIP. Έχει να κάνει με διάφορα πρότυπα, έχει να κάνει με συμβατότητα, έχει να κάνει με προτιμησιακό καθεστώς. Τι σημαίνει αυτό το in particular, το ειδικότερο για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τώρα, για τις υπηρεσίες λέμε ότι η ρήτρα αυτή ισχύει μόνο για τις, για τις μη διακρίσεις. Είναι αυτή η διαπραγματευτική σας θέση. Θα υπάρχει στο κείμενο ή θα εμφανιστεί στο τέλος. Και κυρίως ε, κάτι σημαντικό. Στο ψήφισμα μας λέμε ξεκάθαρα ότι θέλουμε μία συμφωνία που να καλύπτει και το ομοσπονδιακό επίπεδο και το υπο-ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτό το ε, υιοθετείτε στην έκθεσή σας, αλλά προφορικά δεν μας είπατε τίποτα στις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις για το θέμα αυτό. Και για την αηφορία, το σχετικό κεφάλαιο. Ναι, είναι ένα θαυμάσιο κεφάλαιο αυτό που προτείνεται. Όμως λείπει το κομμάτι της θέσης σε ισχύ όλων αυτών. Πότε θα μας τα παρουσιάσετε αυτά, τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν δηλαδή και ε, πώς ακριβώς, ποιο είναι το περιεχόμενο του σχεδίου για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Είναι σαφές το προαπαιτούμενο στο δικό μας ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η διατύπωση είναι αρκετά ασαφής θα έλεγα. οι εταιρείε υποχρεούνται να εμείνουν στι κατευθυντήριε γραμμέ του ΟΣΑ. Και αυτό ήταν ένα από τα βασικά μα προαπαιτούμενα. Θα μπορούσατε και αυτό να το σχολιάσετε. Και τέλο. Κάτι το σημαντικό για το Κοινοβούλιο είναι η κοινοβουλευτική διάσταση όλου αυτού του εγχειρήματο. Στην διαπραγματευτική διαδικασία αυτό το αναφέρατε. Ποιο καθεστώς έχει η κοινοβουλευτική διάσταση στις διαπραγματεύσεις. Και θα δώσω το λόγο τώρα και στους λοιπούς σκιώδεις εισηγητές. Πρώτον η αίμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι έλαβε υπόψη της το ρόλο που θα παίξουμε εμείς σε αυτή τη διαπραγματευτική διαδικασία και είναι αυτό σημαντικό. Κάποια από τα πράγματα στην έκθεση έχουν αλλάξει γιατί έχουν υπάρξει εξελίξεις. Καλό θα ήταν να έχει γίνει αυτή η συζήτηση νωρίτερα. Έστω όμως γίνεται και ακόμα και σήμερα. Πολλά έχουν ήδη υποθεί για την έκθεση. θα πρέπει να έχουμε μια φιλόδοξη και συνολική συμφωνία. Δεν θα υποκύψουμε σε ε, κάποια ρύθμιση επιμέρους μόνο θεμάτων ε, να πάρουμε κάποιες μικρές συμφωνίες ε, που μας προσφέρουν οι, Ευρωπα... οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να είναι συνολική συμφωνία. Παραμένει προτεραιότητα το θέμα των δημοσίων προμηθειών ή αγορών. Είναι απαραίτητο για να υπάρξει συνολική συμφωνία. Ως προς τις γεωγραφικές ενδείξεις, σύμφωνα με τις αναφορές, η διαπραγμάτευση έχει βρεθεί σε τέλμα για το θέμα αυτό. Πώς θα προχωρήσουμε θα συζητήσουμε για την ύπαρξη ενδεχομένω ε, συστήματο εμπορικών σημάτων, trademark, αντί για γεωγραφικές ενδείξει, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση σα συγχαίρω π.χ. για τη δουλειά ε, που έχετε κάνει στο κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πολιτική μου ομάδα και η διαδικτυακή επίλη ε, θα λειτουργήσει ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για όλους όσοι θα, όσοι θα ήθελαν να εξάγουν τα προϊόντα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστώ. Χαίρομαι γιατί συζητούμε για την TTIP και βλέπουμε ότι υπάρχει συνένεση. Είπα και ε, ε. Δεν θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία early harvest. Ε, και αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίσουμε εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Πρόεδρου των ΗΠΑ και άλλων προσωπικότητων. Ε, στις 21 Προελίων αναπετώμε. Εγώ διαφοροποιούμε κάπως από τους συναδέλφους γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό πράγματι να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει υπόψη της αυτό το ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Όμως το ψήφισμα αυτό δεν ήταν το ιδανικό Όλοι συμβιβάστηκαν, επομένως δεν θεωρώ ότι το ψήσμα είναι βίβλος. Εκφράζονται, και Ευαγγέλιο, ε, ε, εκφράζονται φόβοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένος για διάφορα θέματα και αυτό που μου ανησυχεί είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες π.χ. για την πρόσβαση στις αγορές ειδικότερα στο θέμα των δημοσίων αγορών. Είναι βασικό για την Ευρώπη και δεν θα πρέπει οι προτεραιότητες μας να επισκιαστούν ε, και αντί αυτού να ασχολούμαστε με το να τραβούμε κόκκινες γραμμές στην άμμο. Οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλέ, τα αιτήματα είναι πολύ επιτακτικά και από την άλλη δεν υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης γιατί έχουν τραβηχτεί τόσες πολλές κόκκινες γραμμές ταυτόχρονα. Ε, θέλω να μάθω περισσότερα για την πρόσβαση στις αγορές. Χαίρομαι με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη συνάντηση μου με την Greenpeace την περασμένη εβδομάδα προέκυψε ένα ερώτημα και σημειώνω κάτι γιατί ισχύει όχι μόνο για την Greenpeace αλλά και με άλλες ΜΚΟ και με πολίτες με τους οποίους συνομιλώ. Ανησυχούν τι σημαίνει κανονιστική συνεργασία, συνεργασία για κανονιστικά θέματα. Θα παρακαμφθεί έτσι η νομοπαρασκευαστική διαδικασία στα Εθνικά Κοινοβούλια, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε δημοκρατικώς εκλεγμένα όργανα και σε ρετούς εκπροσώπους. Είναι ένας τρόπος να παρακαυθούν όλα αυτά. Τι ακριβώς σημαίνει ε, αυτό ε, ε, κανονιστική συνεργασία και τι ακριβώς δεν σημαίνει και τι είδους ε, ε, συνεργασία διαμορφώνουμε για το μέλλον σε θέματα κανονιστικά, ρυθμιστικά και πώς ακριβώς διαφυλάτετε εσείς το ευρωπαϊκό δικαίωμα του νομοθετή. Ο Χέλμοντ. Thank you, Bernd. As rapporteur. Ευχαριστώ, Μπέντ. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου γιατί τουλάχιστον μπορούμε να μιλήσουμε για την παρακολούθηση, να πούμε πώς έχουν τα πράγματα στις διαπραγματεύσεις μέχρι τώρα και να λάβουμε υπόψη μας και τη θέση του Κοινοβουλίου. Είμαστε κάπου στα μέσα της όλης διαπραγμάτευσης, όπως είπες και εσύ. Σίγουρα λοιπόν υπάρχουν κάποια ερωτήματα ακόμα και κάποιες παρατηρήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο μέχρι δηλαδή τη στιγμή που θα μπορέσουμε να δούμε το όλο κείμενο της συμφωνίας TTIP όπως έχει προχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα να θίξω κάποια σημεία. Υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά απώλειες θέσεων απασχόλησης. Ιδιαίτερα αν παρακολουθήσει κανείς κάποια από τα σημεία τα οποία δεν έχουν ε, επεξεργαστεί. Έχουμε ζητήσει από την Επιτροπή να κάνει μία εις ανάλυση για το κάθε διαφορετικό κράτος μέλος όσον αφορά τις ε, εξελίξεις και στους προσανατολισμούς ε, σε θέματα ανταγωνιστικότητας και βεβαίως τις πιθανές επιπτώσεις όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης. Δεν βλέπουμε αυτό το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Και εδώ θα πρέπει να επιταχυνθεί λίγο η διαδικασία, γι' αυτό και εμείς ασκούμε πίεση. Είναι υποχρέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Υπήρξε επίσης και μια κοινή επιστολή στον αφορά τον αποκλεισμό, την εξαίρεση των ε, δημόσιων ε, υπηρεσιών και δεν βλέπω ούτε στο σημείο 2β7 να αποκλείονται αυτές οι υπηρεσίες ούτε αυτές του γενικού οικονομικού γενικής οικονομικής ε, ωφέλειας. Δεν βλέπω πουθενά να υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις και αυτό και σε σχέση με τη Συμφωνία Τίζα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αυτό είναι ένα περίπου θέμα και πρέπει να το εξετάσουμε. Το θέμα τώρα των προσωπικών δεδομένων και εδώ θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και οριζόντια βασιζόμενη στο άρθρο 14 του συστήματος ε, γενικών προτιμήσεων και σε κάθε περίπτωση εδώ θα πρέπει να συμπεριληφθούν αυτά τα δεδομένα το θέμα των δεδομένων, εν σίγουρα θα επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή δεν τα έχετε επεξεργαστεί. Το 2 Δ 2, σημείο 2 Δ 2, για την ε, έγκριση, υλοποίηση, κύρωση καθώς και όλες τις συμφωνίες που αφορούν τις επιπτώσεις για το περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιστήσουμε για άλλη μια φορά την προσοχή της Επιτροπής σε αυτά τα σημεία τα οποία κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την άποψή μας είναι εξαιρετικά σημαντικά για την βιώσιμη ανάπτυξη και όλο το κεφάλαιο που αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ολοκληρώνω το Κοινοβούλιο. Ζήτησε ένα νέο σύστημα όσον αφορά το θέμα των, της επίλυσης των διαφορών του ISDS. Βεβαίως, τα δικαστήρια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των ΗΠΑ ε, σίγουρα δεν μπορεί να θεωρήσουν ότι υπερτερούν τα προσωπικά ή τα ιδιωτικά συμφέροντα σε σχέση με αυτά των κρατών. Προς το παρόν, λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε αν θα αντικατασταθεί αυτός ο μηχανισμός από έναν άλλον, από τη στιγμή που δεν ξέρουμε ποια είναι η διαπραγμάτευση και το περιεχόμενό της, δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει ένα νέο σύστημα αν θα υπάρξει ένας νέος τρόπος επίλυσης των διαφορών, αν θα παραμείνουμε στον αρχικό. Εμείς πάντως επιμένουμε πρέπει να αλλάξει η λογική αυτού του μηχανισμού επίλυσης των διαφορών του ISDS και όχι να γίνουν απλώς κάποιες διακοσμητικές αλλαγές. Τελειώνω, τελειώνω. Ναι, έτσι τουλάχιστον δεν πρέπει εγώ να επαναλάβω όλα αυτά που είπες σε σχέση με την ε, αξιολόγηση, μελέτη δικτύπου, καθώς και το θέμα του δεσμευτικού χαρακτήρα του κεφαλαίου που αφορά την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Ουσιαστικά εσείς τι κάνετε. Παίρνετε το κείμενο του Κοινοβουλίου, αλλά δεν είναι δεσμευτικό το κείμενο που προτείνετε. Δηλαδή το ρήμα shall γίνεται may στα αγγλικά και βλέπουμε ότι με μια τέτοια αλλαγή αλλάζει τελείως η ισχύ του κειμένου. Τώρα, όσον αφορά δασμολογικές ποσοστώσεις, μιλάμε για 300.000 τόνους για το χείριο κρέας ή για το βόλιο κρέας. Ο κύριος Δεμαρτή μας είπε ότι είναι μόνο το 1 ή το 2% της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, ξέχασε μάλλον αν και ήταν πρώην ε, για θέματα γεωργίας, πώς λειτουργεί το θέμα της ελαστικότητας και ότι αυτό το 1 ή 2% μπορεί να επηρεάσει και τα έσοδα των ε, γεωργών αλλά και τις τιμές. Θα ήθελα λοιπόν να μας πει ακριβώς για το χερνό αλλά και για το βόλιο κρέας πώς ακριβώς βλέπει την επίπτωση για αυτές τις ε, ποσότητες μας μίλησε και για τη σχέση μεταξύ TISA και TTIP. Πώς ακριβώς λαμβάνετε υπόψη σας το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ΤΙΖΑ, και για τους καταλόγους και για τις ρήτρα για το status quo παραδείγματο χάρη. Πώς βλέπετε τη διασύνδεση συγκεκριμένα εσείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ TISA και TTIP και βεβαίως για το ICS που για μένα είναι ISDS, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αν κατάλαβα καλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το ICS ουσιαστικά δεν είναι στο μεικτό τμήμα της συμφωνίας, αλλά είναι θέμα ευρωπαϊκής αρμοδιότητας. Ποια είναι λοιπόν η επίσημη θέση της Επιτροπής για το θέμα αυτό, για το καθεστώς του ICS. Αν διαπραγματεύεστε, διαπραγματεύεστε, συγγνώμη, εδώ το ίδιο με αυτό που διαπραγματεύεστε με την ε, ΣΕΤΑ, μπορεί να υπάρξει πριν τις εθνικές κυρώσεις, μετά δηλαδή την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μία προσωρινή θέση ισχύ του ΣΥΤΑ. Και βλέπει κανείς ότι το ICS θα αρχίσει να ισχύει για τρία χρόνια ακόμα και στις χώρες αυτές που δεν δέχονται την τελική συμφωνία, που δεν θα κυρώσουν δηλαδή την συμφωνία ΣΕΤΑ. Ακόμα δηλαδή και σε αυτή τη χώρα μπορεί να υπάρξει προσφυγή κατά του κράτους αυτού επί τρία χρόνια. Αν λοιπόν όντως διαπραγματεύεστε το ίδιο πράγμα με τις ε, ε, Ηνωμένες Πολιτείες, και αν πρόκειται για αρμοδιότητα ευρωπαϊκή θέλουμε να το ξέρουμε εμείς ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σαρνέζ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλα αυτά τα θέματα που έθιξαν οι συνάδελφοι δείχνουν ότι όντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη σε αυτά που ψηφίζει και αυτά που επιθυμεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει. Και καταλαβαίνετε ότι αν εμείς ε, τοποθετούμαστε για κάποια θέματα και οι διαπραγματευτές που διαπραγματεύεται εξ ονόμα Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λαμβάνουν υπόψη αυτές τις θέσεις, εμείς πραγματικά ανησυχούμε. Είναι μάλιστα και αντιδημοκρατικό. Είπατε ότι ελπίζετε να υπάρξει εντολή πριν το τέλος της Προεδρίας Ομπάμα. Μα καμία πιθανότητα δεν υπάρχει τόσο χρόνο διαπραγματεύεστε. Αλλά από τη στιγμή που πέρασε το δικό μας ψήφισμα, είδαμε ότι αυτά που λένε οι υποψήφοι και οι δημοκρά... του Δημοκρατικού αλλά και του Ρεπουμπλικανικού κόμματος και η Χίλαρη Κλίντον και ο υποψήφιος του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων έχουν εκφράσει πολλές πολλές επιφυλάξεις έναντι αυτής της εμπορική συμφωνίας και όσον αφορά τη μείωση της απασχόλησης, έλλειψη διαφάνειας. Βλέπετε ότι τελικά και οι Αμερικανοί και εμείς λέμε ίσως κάποια κοινά πράγματα. Μήπως θα πρέπει να βγείτε λοιπόν από την διαπραγμάτευσή σας και να ακούσετε τι λέμε. Ο Γιάννη Ζαντό μίλησε και για το μεικτό χαρακτήρα αυτής της σύμβασης. Είναι θέμα δημοκρατίας και επί μήνες δεν μπορούμε να ακούμε ναι είναι, δεν είναι μεικτή συμφωνία. Καλό θα ήταν να το ακούσουμε, να το δεχτούμε και να δούμε αν ναι ή όχι αυτή η προσωρινή ισχύς, ισχύ, ακομα και αν μια χώρα απορρίψει και δεν κυρώσει ποτέ τη συμφωνία. Θα ήθελα λοιπόν να μας απαντήσει η Επιτροπή. Τα λέω και τα ξαναλέω αυτά, δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούτε, αλλά φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προσέχει και δεν απαντάει. Το θέμα μου είναι πάντα και εκ νέου το θέμα των κρατικών προμηθειών. Το 90% αν θέλετε των ε, ευρωπαϊκών ε, αγορών είναι ανοιχτά όταν πρόκειται για τέτοιες δημόσιες προμήθειες. Οι Ηνωμένε Πολιτείε αντίθετα προστατεύουν την αγορά τους και προσπαθούν να βοηθήσουν πολύ περισσότερο τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θα έπρεπε λοιπόν ίσω και εμεί να το δούμε αυτό, να εμπνευστούμε και να δημιουργήσουμε ένα Small Business Act στην Ευρώπη. Τζουντ. Συμμερίζομαι τη δική σας ανησυχία Εάν η Επιτροπή δεν ανταποκριθεί στην, στην έκθεση συγγνώμη, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα μας ε, φέρει κάτι τέτοιο σε δινή θέση. Και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου θα ερχόταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας εκδημοκρατισμός υπό την έννοια του ελέγχου των εμπορικών πολιτικών. Θα πρέπει να ανταποκριθεί η Επιτροπή και σε αυτό. Με βάση τις ανησυχίες ε, του Κοινοβουλίου ήθελα καταρχήν να πω για το TTIP ότι έχει επιτελεστεί πρόοδος σε σχέση με δημοκρατικό έλεγχο, διαφάνεια και ούτω καθεξής. Πολλά έχουν γίνει, ιδιαίτερα για τη διαφάνεια, αλλά με μια τέτοια έκθεση τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί αν δούμε ένα από τα ζητήματα κλειδιά στην Επιτροπή μας, θα αφορούσε τον αποκλεισμό δέκο, ιδιαίτερα δέκο, από πλευράς Επιτροπής. Η Επιτροπή λέει ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα σε σχέση με τις υπηρεσίες δημόσιου συμφέροντος. Εμείς δεν παίρνουμε θέση για να πάρουμε θέση και μόνο. Οι δημόσιες υπηρεσίες της ε, εμπορικές συμφωνίες έχουν ε, φυγεί με βάση τους ε, χρήστες και τους δημόσιους φορείς. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να δούμε τις ενδυνάμει επιπτώσεις μιας επίλυσης διαφοράς. Είτε πρόκειται για κράτος επενδυτή είτε όχι. Τώρα, στην Επιτροπή Ίντα υπήρξε ομοφωνία. και δεν τροποποιήθηκε στην Ολομέλεια η έκθεση αυτή. Δηλαδή, έτυχε ευρεία συνένεση. Όμως η Επιτροπή τι μας λέει, εμείς δεν θα αλλάξουμε αυτό που κάνουμε στις εμπορικές μας διαπραγματεύσεις. Όλα έχουν ε, καλώς. Κοιτάξτε προς άλλη κατεύθυνση. Υπάρχει όμως πρόβλημα. Εάν δεν γίνουν αλλαγές στην διαπραγμάτευση, τότε εμείς θα ασκήσουμε το δικαίωμα αρνησικυρίας και θα ήταν τρομερό να σας το έχουμε θίξει εκ των προτέρων γιατί μιλάμε για την εμπιστοσύνη του κοινού. Και η Επιτροπή Περιφερειών το έχει θίξει και η ΕΟΚΕ. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δώσετε περισσότερες εξηγήσει από αυτά που βλέπουμε στην ε, έκθεση, γιατί η πρόοδος που επιτελείται αφορά την επανάκτηση της εμπιστοσύνης του κοινού και έτσι θα τη Θα ήθελα να η Επιτροπή να ανταποκριθεί λίγο καλύτερα στη θέση του Κοινοβουλίου. Κάρολιν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κάτι σε σχέση με αυτό που μόλις είπε η Τζουδίχα Είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τους ε, εκπροσώπους του κλάδου από την Αμερική και έχω την εντύπωση ότι η στάση τους ήταν πολύ θετική, τουλάχιστον από αυτά που ακούσαμε. Αυτό που μας ε, είπαν είναι ότι από μέρος τους είναι κάπως απογοητευμένοι γιατί θεωρούν ότι από τη στιγμή που κοιτάμε να πετύχουμε τον ίδιο στόχο είναι πάρα πολύ κρίμα που οι παρατηρήσεις και τα μηνύματα που βγαίνουν προς τα έξω είναι σχετικά αρνητικά και ότι από τη στιγμή που οι Ηνωμένε Πολιτείε δέχτηκαν κάποιες από τις μας προτάσεις και υποχώρησαν και έγιναν σωστά βήματα τουλάχιστον προς τη σωστή κατεύθυνση συνεχίζουμε να αναφερόμαστε σε αυτά που δεν πάνε καλά. Μιλάμε για λήψη διαφάνειας, το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η στάση δεν εμπνέει καθόλου τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι δέχομαι αυτά που είπε η Τζούντ. Το ψήφισμα δεν είναι βίβλος, αλλά εκπροσωπεί τη μεγάλη πλειοψηφία που εκφράστηκε στο Κοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε συνεπείς, να ζητήσουμε από την Επιτροπή να ενσωματώσει ορισμένα στοιχεία που ανέφερε μια μεγάλη πολιτική πλειοψηφία. Διαφορετικά τι νόημα έχει εκ των υστέρων μετά τη διαπραγμάτευση να ψηφίσουμε υπέρ ή κατά. Τότε θα περιοριζόμασταν κοινοβουλευτικά. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε με την επιρροή μας. Για παράδειγμα, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και οι μεγαλύτεροι, περισσότεροι φορείς λένε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη της ΜΜΕ σε αυτή την ε, συμφωνία ελευθέρου εμπορίου. Λέμε ότι οι ΜΜΕ είναι σημαντικές. Όταν όμως δούμε το κείμενο υποδιαπραγμάτευση βλέπουμε ότι το κεφάλαιο αυτό δεν είναι δεσμευτικό και δεν λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες των επιχειρήσεων, διότι το 62% των ΜΜΕ της Γερμανίας είπαν ότι αντιτάσσονται στο TTIP. Δεν το κάνουν για ιδεολογικούς λόγους, το κάνουν γιατί δεν ε, βρίσκουν να αντικατοπτρίζεται η θέση τους. Έπειτα το δικαίωμα ρύθμισης. Αν έχουμε την, ε, ε, το κανονιστικό πλαίσιο και το ICS από την άλλη, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Η Επίτροπη λέει ε, δηλώνω το δικαίωμα ρύθμισης, αλλά πώς το θέτει σε εφαρμογή. Γιατί αν διαβάσουμε το κείμενο βλέπουμε ότι υπάρχει αποδυνάμωση. Επίσης, σε σχέση με τα ε, πρότυπα, της προδιαγραφές του περιβάλλοντος και της εργασίας, θα θέλαμε να αναφέρονται σε όλα τα κεφάλαια και δεσμευτικά. Σήμερα είναι διαφορετικό το πλαίσιο αναφέρονται σε ένα κεφάλαιο το οποίο δεν είναι δεσμευτικό. Όπως είπε και η Τζούντ, έχουμε το δηλωτικό σκέλος, το οποίο αποτελεί το καλό μάρκετινγκ της Επιτροπής, αλλά υπάρχει και ο αντίποδας που δεν λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσει του ψηφίσματος. Αυτή είναι μια προειδοποίηση για την Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Σάντρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ανήκω σε αυτούς που ζητούν περισσότερες διευκρινήσεις για το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. Να πω ότι υπάρχουν εργασιακά πρότυπα, δεν πρέπει να χαμηλώσουν αυτά, όμως δεν γίνεται αναφορά στη σύμβαση, κυρίως ως προς τη Γεωργία, τους αγρότες και αυτά. Και τα περιβαλλοντικά πρότυπα τι εννοεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς όταν αναφέρεται στην αρχή της προφύλαξης. Πρέπει να μας δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Και τρίτον, δεν είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος με τις πληροφορίες που μας δώσατε. Από τη μία μας λέτε δεν απειλούνται οι γεωγραφικές ενδείξεις, όλα καλά πάνε. Και από την άλλη μας λέτε δεν έχουν προχωρήσει διαπραγματεύσεις ε, ως προς αυτό. Όταν ζητούμε δηλαδή περισσότερες διευκρινήσεις, αυτό μας απαντάτε. Και από την άλλη αναφέρεστε στο ότι θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Με ανησυχεί αυτό που μας λέτε. Θα ήθελε η Επιτροπή να μας πει συγκεκριμένα με γεγονότα, με περιστατικά που βρισκόμαστε σήμερα σε, ως προς τη διαπραγμάτευση για αυτά τα τρία θέματα. Και Παρακολουθούμε όλη την προεκλογική εκστρατεία στη ΣΥΠΑ. Συνεχίζουμε ε, να διαπραγματευόμαστε χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τι λέει ο κάθε υποψήφιος ή ε, συμπεριλαμβάνουμε στη διαπραγματευτική μας στρατηγική τα γεωπολιτικά στοιχεία που προκύπτουν νομίζω ότι δεν είναι υπεύθυνο και πολιτικός είναι επικίνδυνο να μην λάβουμε υπόψη την κατάσταση έτσι όπως εξελίξεται στην προεκλογική εκστρατεία σήμερα στη ΣΥΠΑ. Ευχαριστώ, η Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής σας για τις πολύ έγκυρες ερωτήσεις τους, οι οποίες απτώνται πολλών και διαφορετικών θεμάτων και θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο πιο συγκεκριμένα μπορώ στα σχόλιά σας. Επιτρέψτε μου όμως να πω καταρχάς το εξής. Στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου εμείς θα, ε, δεν φιδόμαστε προ, προσπαθειών έτσι ώστε η συμφωνία αυτή να ταιριάζει ώστε να το περισσότερο με την εντολή που μας έχετε δώσει. Και είμαστε αρκετά έξυπνοι ώστε να γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε τη στήριξη του Κοινοβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, έναντι του Συμβουλίου βέβαια. Τώρα, αν παραμένουμε, ε, παραμένουν ερωτήματα τα οποία δεν σας ικανοποιούν, τότε θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά και ατομικά θα έλεγα Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βουλευτές, έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις. Θα έλεγα όμως το εξής. Διαπραγματευόμαστε με ένα πολύ ισχυρό εμπορικό εταίρο που έχει αναλάβει ηγετική θέση στους διεθνείς κανόνες εμπορίου τα τελευταία 50 και 60 χρόνια. Επομένως είναι δύσκολη η διαδικασία αυτή είτε συνδέεται με θέματα που μας αφορούν επιθετικά είτε συνδέεται με θέματα που μας αφορούν αμυντικά. Είμαστε μέσω διαπραγμάτευσης, σας υπενθυμίζω, και δεν είναι αυτή πάντοτε εύκολη. εύκολη. Έχουμε δηλαδή μονίμως ε, τετρακίνηση ε, επιλέξει στο κυβότιο των ταχυτήτων, στο όχημα που οδηγούμε. Και ισχύει αυτό και για τους Αμερικανούς ε, ο ομολόγος μας και εταίρους μας. Να ξεκινήσουμε με τις δικές σας ε, ερωτήσεις κύριε Πρόεδρε για το επίπεδο καλής διαβίωσης των ε, ζώων. Στο κεφάλαιο SPS έχουμε κάνει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Οι απόψεις μας είναι σαφής. Αν δείτε την καταστατική προσέγγιση για την καλή διαβίωση των ζώων θα το κατληφθείτε αυτό. Πρέπει να φτάσουμε σε συμβιβασμό γιατί η καταστατική προσέγγιση των Αμερικανών είναι διαφορετική όμως η πρόταση που έχουμε εμείς κάνει θεωρούμε ότι συνάδει πλήρως με το μέλημα αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και άλλων Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καλή διαβίωση των ζώων και τα σχετικά πρότυπα. Και η Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος ε, ε, ενδιαφέρεται ιδιαίτερως για το θέμα αυτό. Τώρα ως προς τα προσωπικά δεδομένα, το άρθρο 14 και το ΚΑΤΣ. Το μόνο πάνω στο οποίο μπορώ να δεσμευτώ αυτή τη στιγμή είναι ότι εμείς θα προστατεύσουμε πλήρως, να ε, προστατεύσουμε, θα προστατεύσουμε πλήρως την προσέγγιση ε, της προστασίας των δεδομένων, της προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας έτσι όπως την έχουμε ορίσει εγχωρίως στην Ευρώπη και με τη συνθήκη της Λισαβόνας και με άλλα κείμενά μας. και θέλουμε όλα αυτά να ε, ε, απεικονιστούν στη διαπραγμάτευση και στη συμφωνία με τους Αμερικανούς εταίρους και φίλους μας. Τώρα, όταν κανείς διαπραγματεύεται μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, ε, καταρχήν η διαπραγμάτευση γίνεται μεταξύ των δύο συμβαλόμενων μερών στην εκάστοτε συμφωνία και αυτό αποκλίνει από την προσέγγιση του ΠΟΕ. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά προσπαθούμε τα κανονιστικά και ρυθμιστικά μας συστήματα να τα κάνουμε πιο συμβατά μεταξύ τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της συμμόρφωσης με τους νόμους σήμερα είναι κατά μέσο όρο υψηλότερο για μια επιχείρηση από ότι είναι το κόστος πληρωμής του δασμού για την εκάστοτε εισαγωγή. Με δεδομένο λοιπόν αυτό, οτιδήποτε γίνει για τη μείωση μη απαραίτητων μη απαραίτητου κόστου συμμόρφωσης με νομοθεσία είναι καλό πράγμα και υπογραμμίζω ε, την, ε, τον επιθετικό προσδιορισμό μη απαραίτητου ε, κόστου συμμόρφωσης με την ε, νομοθεσία. Το μη απαραίτητο υπογραμμίζω και αυτό βεβαίως πάντοτε ωφελεί και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και οι ανεξάρτητες μελέτες και έρευνές μας το έχουν αυτό αναδείξει ξεκάθαρα. Στις δημόσιες αγορές το προτιμησιακό καθεστώς σίγουρα έχει μεγάλη επιρροή και σε επίπεδο πολιτείας ή και σε επίπεδο χαμηλότερο από την πολιτεία, όχι μόνο σε μοσπονδιακό, θα είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αυτό, αλλά και σε πολλούς Τομεί στα επαγγελματικά προσόντα ε, διέπονται από νομοθεσία που ορίζεται σε υπο-ομοσπονδιακό επίπεδο και εμεί θέλουμε ένα μηχανισμό για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνομιλήσουμε και με εταίρους ε, σε επίπεδο κάτω του ομοσπονδιακού, σε επίπεδο πολιτείας. Καθώς προχωρούμε με τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής στο χρηματοπιστωτικό τομέα, ε, σίγουρα πρέπει να εξετάσουμε την ομοσπονδιακή διάσταση όλων αυτών για τη θέση σε ισχύ και εφαρμογή του κεφαλαίου για τα εργασιακά και το περιβάλλον. Πολύ λογική και θεμητή η ερώτησή σας. Τι μπορώ να πω γι' αυτό. Ε, στις παρελθούσες εμπορικές συμφωνίες τι έχουμε δει. Οι ΙΠΑ επιβάλλουν εμπορικές και χρηματοοικονομικές κυρώσεις για να εφαρμόσουν τις συμφωνίες που έχουν συνάψει. Εμείς δεν έχουμε φτάσει στο απότατο σημείο στο οποίο θα εφαρμόζουμε εμπορικές κυρώσεις, ποινές δηλαδή και ε, χρηματοοικονομικές. Θέλουμε να συμφωνήσουμε πρώτα με τους Αμερικανούς για το είδος των δεσμεύσεων στις οποίες θέλουμε να καταλέξουμε μαζί για το περιβάλλον και για τα εργασιακά, διότι σε αυτό το στάδιο πρέπει να ασκήσουμε ηγεσία, να δείξουμε τι σημαίνει τον 21ο αιώνα μια συμφωνία που εμπνέεται από αρχές και εμπνέει αρχές πέρα από το άνοιγμα το απλό των αγορών. Και στη συνέχεια με τους ομολόγους μας θα είμαστε σε θέση να αποφασίσουμε μαζί ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό μοντέλο για να διασφαλίσουμε την πλήρη συμμόρφωση ε, στα προβλεπόμενα από τη συμφωνία. Άπαξ και ακυρωθεί η TTIP, θέλουμε και φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και από την Αμερικανική πλευρά, το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλακεί πλήρως στη θέσπιση των προτεραιοτήτων και των επιμέρους στόχων της διατλαντικής εργασίας που πρέπει να φέρουμε σε, πέρος, σε πέρας. Βεβαίως δεν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό λήψης απόφασης παρά το κοινοβούλιο ή παρά τα ε, ε, κοινοβούλια ε, και το συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Και όποια προσέγγιση και αν πάνω σε όποια προσέγγιση και αν και συμφωνήσουμε με τους Αμερικανούς ομολόγους μας, η διαδικασία θα είναι η γνωστή που θα ακολουθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ελπίζω αυτό να σας καθησυχάζει. Τώρα ως προς τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τη φιλοδοξία. Ναι, θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι, αλλά δεν σας κρύβω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι των διαπραγματεύσεων που έχει να κάνει με την πρόσβαση στην αγορά. Δουλεύουμε για να βρούμε έναν τρόπο να υπάρξει το μήνα, παροχωρήσουμε για τα θέματα των δημοσίων αγορών, για τις υπηρεσίες, για τη γεωργία, για τις γεωγραφικές ενδείξεις, για τις βασικές αυτές συνιστώσεις ε, που θα διαμορφώσουν την τελική συμφωνία και την εικόνα αυτής. Όμως νομίζω ότι είναι ευρέως γνωστό το ότι έχουμε δει ότι οι διαπραγματεύσεις για το τελευταίο 3% των δασμολογικών γραμμών που είναι και ε, οι πιο ευαίσθητες ε, για εμάς θα γίνουν στο τέλος. Όταν μας ρωτούν αν ήδη μιλάμε για ποσότητες με τους Αμερικανούς ομολόγους μας απαντούμε όχι, τουλάχιστον εγώ δεν το γνωρίζω, γιατί είναι κάτι που έχουμε σαφέστατα αφήσει για το τελικό ε, στάδιο των διαπραγματεύσεων. Δεν θα σας κρύψω ότι η πρόοδος για τις δημόσιες αγορές και τις γεωγραφικές ενδείξεις τους τελευταίους δύο μήνες έχει σημειωθεί με πάρα πολύ αργά βήματα και θα πρέπει να υπερπηδηθούν διάφορα εμπόδια για το θέμα αυτό ε, πριν ξεκινήσει το endgame, το τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων. Ίσως σε αυτό μπούμε το καλοκαίρι, έτσι αφήνουν να εννοηθεί οι Αμερικανοί, εάν έχουμε ένα κείμενο ε, που να αφορά σε όλες τις διαπραγματεύσεις. Ίσως το τελικό στάδιο δηλαδή ξεκινήσει το ε, καλοκαίρι. Τώρα είμαστε στο μεσαίο στάδιο, δεν είμαστε στο endgame, είμαστε στο middle game. Και πρέπει να βρούμε τρόπους να χτίσουμε, ε, να δομήσουμε καλύτερα το παιχνίδι σε αυτό το μεσαίο στάδιο πριν μπούμε ε, στη συζήτηση για τις δημόσιες αγορές. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το συζητήσει αυτό εσωτερικά την Παρασκευή. Κύριε Σούλτς για το θέμα των επιπτώσεων στις θέσεις απασχόλησης, ε, μια συμφωνία σαν την TTIP. Πράγματι, εμπορικές συμφωνίες, κάθε εμπορική συμφωνία έχει ε, ε, αντίκτυπο στις θέσεις απασχόλησης ε, προς όλες τις κατευθύνσεις, ορισμένοι κλάδοι της οικονομίας κερδίζουν, άλλοι χάνουν. Θεωρούμε ότι είναι θετικό το γενικό πρόσημο και θα είναι θετικό το γενικό πρόσημο. Σε έξι εβδομάδες θα γίνει, θα δημοσιευθεί η προσωρινή έκθεση για την ε, ε, αηφορία, τη βιωσιμότητα. Είναι μια ανεξάρτητη έκθεση που θα υποβληθεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 4 με έξι εβδομάδες. Τώρα για τις δημόσιες υπηρεσίες. Εκτός και αν προτείνει κάποιος ότι έχουμε υπάρξει αυτά αρέσκη, θα ήθελα να πω ότι μας έχει απασχολήσει πολύ το θέμα τελευταία. Όλη αυτή τη χρονιά έχουμε δουλέψει εντατικά. Δημόσια δήλωση υπήρξε από πλευράς ε, ε, Επιτρόπου. Είχαμε ε, πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις σε επίπεδο RSDR και έχουμε τέσσερα firewall, τέσσερις τείχους προστασίας στις προτάσεις που έχουμε υποβάλει προς τη ΣΥΠΑ. Ευρύτερη καταρχάς εξαίρεση των δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πεδίο της ε, ε, κυβερνητικής αρμοδιότητας, παράρτημα 2 επιφυλάξεις που είναι εξαιρετικά ευρείες στο ε, θέμα των υπηρεσιών και της παροχής αυτών, αλλά βεβαίως οποιοδήποτε από εσάς μπορεί να, να τον φέρω σε επαφή με τους εμπειρογνώμονες και τους ειδικού από τις υπηρεσίες μας, γιατί βλέπω ότι δεν έχετε πιστεί και είναι δική μας δουλειά να σας πείσουμε και να σας εξοικειώσουμε με την νομική φύση των επιφυλάξεων για τις δημόσιες υπηρεσίες που έχουμε θέσει στη διαπραγμάτευση και στη συμφωνία αυτή. Βεβαίως η TTIP θα είναι ένα νομικό κείμενο έκτασης 2.000 σελίδων, επομένως η νομική διατύπωση είναι αυτή που θα καθορίσει το βαθμό στον οποίο προστατεύονται οι εκάστοτε κλάδοι της οικονομίας. Όμως, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχουν υπάρξει υποθέσεις επίλυσης των ΠΟΕ ε, διαφορών για θέματα δημοσίων υπηρεσιών και εμείς και οι Αμερικάνοι, οι Αμερικανοί ομόλογοι μας είναι σαφείς στο θέμα αυτό. Δεν θέλουμε η TTIP να περιορίσει τον ε, ζωτικό πολιτικό χώρο για τις κυβερνήσεις να ε, συμπεριλάβουν τις δημόσιες υπηρεσίες μεταγενέστερα. Σημειώνω αυτά που μας είπατε για τη σύμβαση του ε, Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και του ε, συστήματος για την ε, επίλυση διαφορών σε θέματα επενδύσεων από το σχετικό δικαστήριο. Νομίζω ότι αυτά αντέχουν στην πολιτική διοκιμασία, αυτά που προτείναμε είναι δίκαια, είναι διαφανή και συνάδουν με ευρέως και διεθνώς αποδεκτές νομικές ε, διαδικασίες όπως είναι η Χάγη ή το Διεθνές Δικαστήριο Επίλυσης Διαφορών, το ISDS. Άλλωστε ο κύριος Μπράουν σας έχει δείξει ότι εμείς κερδίζουμε όλες σχεδόν τις υποθέσεις και έχουμε και καλύτερο ρεκόρ από ότι οι Αμερικανοί, ε, ο ομόλογοι μας. Ο πρόεδρος διακόπτει και λέει τώρα θα πρέπει να συνεχίσουμε στα αγγλικά γιατί η διερμηνία υπάρχει μέχρι τις 6.30. Ο πρόεδρος ευχαριστεί ευγενικά τους διερμηνείς. Θα σας δω αύριο λέει. Ευχαριστούμε και εμείς. Συνεχίζεται η συνεδρία στα αγγλικά. Uh, ε, Jadot's points about TRQs for beef and pork. We're not there yet. Uh, that is clearly endgame. And when we start talking about those uh, volumes, uh, that is when we will be